Ahora sí. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φιλοξενούμενοι, Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί σήμερα την επέτειο των καλύτερων 60 χρόνων της ιστορίας της ελεύθερης Ευρώπης. Αυτή η στιγμή πρέπει να μας θυμίσει ότι όχι, και να μας θυμίσει όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα ότι οι πολίτες, οι πολίτες είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης περιπέτειας της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Χωρίς τους λαούς της η Ευρώπη απλούστατα δεν υπάρχει. Η ενέργεια, η δύναμη, η νομιμοποίηση για να δράσει προκύπτει από τη δική μας συμμετοχή ως πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να επανασυνδεθούμε με τους πολίτες. Η Ευρώπη πρέπει να έρθει κοντά στους πολίτες, στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο καθήκον που ανέλαβα όταν ανέλαβα αυτό το αξίωμα. Εμείς, 751 εκλεγμένοι άρχοντες, με την υποστήριξη τόσων καλών υπαλλήλων θα πρέπει να εργαστούμε, ούτω ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μην μείνουν κλειστά σαν φρούρια με κινητές γέφυρες που ρίχνουμε και σηκώνουμε. Θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες, να βγούμε έξω, να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να καταλάβουμε, να βάλουμε τα προβλήματα των πολιτών, την αξιοπρέπεια των ανθρώπων στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Οι πρόσφατες Ολλανδικές εκλογές επιβεβαίωσαν ότι δεν κουραστήκαμε από την Ευρώπη μας. Απλώς θέλουμε να λειτουργήσει καλύτερα. Να επιλύσει τα προβλήματα. Την ανεργία, κυρίως των νέων, τη δρομοκρατία, τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, την προστασία των, γυναικών, δικαιωμάτων των γυναικών, των πιο αδυνάτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο συγκεκριμένη, πιο απτή. Μια Ευρώπη των πράξεων, μια πραγματική Ευρώπη. Αρκεί να έχει κανείς λίγη λογική για να καταλάβει ότι αν αποδυναμώσουμε την Ευρώπη δεν πρόκειται να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Κανένα κράτος μέλος, ακόμα και τα πιο μεγάλα και τα πιο δυνατά, δεν μπορούν από μόνα τους να διαπραγματευτούν με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία ή με την Ινδία. Να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές από την Αφρική τη Μέση Ανατολή, να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντά μας, να σταματήσει τη θέρμανση του πλανήτη, να διατρανώσει τις αξίες με τις οποίες όλοι ταυτιζόμαστε. Σήμερα, περισσότερο παραποτέ, εν τη ενώση ισχύς. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε τις προκλήσεις που μας καραδοκούν, που μας περιμένουν. Αισθάνθηκα προσβεβλημένος, όπως φαντάζομαι και όλοι σας, όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε φασισμούς και ναζισμούς, μιλώντας για κάποιες από τις χώρες μας. Η Ευρώπη είναι ο φάρος στον κόσμο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαστε η μόνη ήπειρος που δεν έχει θανατική ποινή. Είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από μια αγορά και ένα νόμισμα. Είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι και μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να ασκούμε αυτό τον ηγετικό ρόλο και να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες και να παροτρύνουμε τους γείτονές μας να μην διολυστήσουν προς ανελεύθερους εθνικισμούς. Ας συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Και τώρα, με χαρά, σας παρουσιάζω τους δύο προσκεκλητμένους μας. Ο πρώτος προσκεκλημένος είναι η Μπάρμπαρ Χέντριξ. Κατάγεται από την, το Άρκανσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Μπάρμπαρα είναι Σουηδέζα και Ελβετίδα πολίτης. Είναι πρέσβυρα του ΟΗΕ, της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, με τη μεγαλύτερη θητεία. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος Barbara Hendricks για την υγεία και την συμφιλίωση, που συντονίζει τη δουλειά για τους πρόσφυγες και για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Hendricks, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ Έχετε το λόγο. Good morning. Bonjour. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εγκεκριμένοι προσκεκλημένοι, φίλοι τη Ευρώπη, είναι μεγάλη η τιμή του να βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα της ολομέλεια με την ευκαιρία της 60 η επαιτίου της Συνθήκης της Ρώμης. Μου ζητήθηκε να εκφωνήσω το λόγο μου στα αγγλικά και θα συνεχίσω στα αγγλικά. Οι σημαντικές επέτειοι μας εμπνέουν να στρέψουμε το βλέμμα στο δρόμο που έχουμε διανύσει και να αξιολογήσουμε την πρόοδό μας. Μας δίνουν επίσης την ευκαιρία να τιμήσουμε τη διορατικότητα εκείνων που μας έβαλαν σε αυτό το φιλόδοξο ταξίδι. Σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας πρέπει ταυτόχρονα να διαρωτηθούμε πώς θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω για ένα πιο φωτεινό μέλλον. Μια κατάρα λέει να ζεις σε ενδιαφέρουσες εποχές. Και αυτό σημαίνει ε, εποχές φόβου, βίας, ξεσηκωμών. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η εποχή μας είναι γεμάτη από βεβαιότητες, κινδύνους και πολλαπλές κρίσεις. Η αχαλήνωτη απληστία των αδίστακτων χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών θεσμών μέχρι και σήμερα έχει μείνει ατιμόρυτη, έχει προκαλέσει ωστόσο διεθνή οικονομική κρίση με καταστροφικές συνέπειες μια παγκόσμια οικονομία σε εκτροχιασμό, καλπάζουσα ανεργία και άνευ προηγουμένου και επέσχυντο επίπεδο ανισοτήτων και μέτρα λιτότητας που άδικα τιμωρούν τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας. Είμαστε στην ενδεκάτη ώρα μιας κατεπίγουσας οικολογικής κρίσης. Έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος για να σώσουμε τον πλανήτη, αλλά εξακολουθούμε να δηλητηριάζουμε τα νερά της γης, τον αέρα της γης, να οδηγούμε στην εξαφάνιση πολύτιμα είδη της χλωρίδας και της πανίδας η παγκόσμια τρομοκρατία, μια βάρβαρη επιδημία που καθοδηγείται από το μίσος και που κατά ένα βαθμό καθοδηγείται από τους ανήθικους ή τροφοδοτείται από τους ανήθικους και παράνομους πολέμους που έχουν ε, ξεκινήσει στο όνομά μας, στοχεύει αθώους πολίτες σε όλο τον κόσμο και προσπαθεί να μας παρασύρει σε έναν φαύλο κύκλο της βίας. Αύριο θα χαιρετήσουμε με μεγάλη θλίψη θα μνημονεύσουμε τα θύματα της ε, άφρονος επίθεσης στο αεροδρόμιο και εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουν ε, επεκταθεί σε όλη την υφήλιο ε, συγκρούσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει πρωτόγνωρες ανθρωπιστικές κρίσεις. Πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να καταλήψουν τις αιστείες τους. 10 εκατομμύρια είναι απάτριδες. 600.000 από αυτούς ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ύπατη αρμοστία για, για τους ε, πρόσφυγες ποτέ δεν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοιου είδους ε, ε, προβλήματα και τόσο πρωτόγνωρε ο μέγεθος καταστροφής από την ίδρυσή της από το 1951. Όλα τα κράτη-μέλη της ΥΠΑ της Αρμοστίας είναι και συμβαλόμενα στις συμβάσεις για τους πρόσφυγες που όχι μόνο εγγυούνται το δικαίωμα της αναζήτησης ασύλου αλλά έχουν ταυτόχρονα ενσωματώσει και διασφαλιστικές δικλείδες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Όταν το 1954 τον Ιούλ, ε, μάλλον η σύμβαση ετέθησε ισχύ το 1954 τον Ιούλιο, όταν το 1956 τα σοβιετικά τάγκς μπήκαν στην Βουδαπέστη για να σταματήσουν την Ουγγρική Επανάσταση, 200.000 Ούγγροι κατέφυγαν στην Αυστρία. Η ύπατη αρμοστία του αναγνώρισε μια πρία ένα πρίμα φάκι καθεστώ ε, προσφύγων και ηγήθηκε τις προσπάθειες για την επανεγκατάστασή του. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η παρέμβαση ήταν εκείνη που διαμόρφωσε και τους ε, ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις κρίσεις. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε και υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στο Σαν Φρανσίσκο. Εγώ ήμουνα μόλις, 20 ημερών εκείνη τη μέρα. Οι γονείς μου δεν είχαν ιδέα για τη διακήρυξη αυτή, όμως ήξεραν πολύ καλά τι σήμαιναν οι νόμοι Jim Crow, οι νόμοι του Apartheid που χώριζαν τις φυλές στο Νότια Αμερική. Εγώ κατ' ουσία είχα γεννηθεί άπατρες στην ίδια μου τη χώρα. Δεν μπορούσα να έχω την ίδια προστασία που προσφέρει ο νόμος, ούτε τα ίδια αναπαλωτρία τα δικαιώματα, γιατί γεννήθηκα κορίτσι στο Στίβενς του Άρκανσο. Ε, παιδί έγινα μάρτυρα των κινημάτων για τα ατομικά δικαιώματα, της προσπάθειας της Ταραλέας Ρόζα Πάρξ και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και όταν υπεγράφει ο νόμος για την καθολική ψηφοφορία το 1964 τον Ιούλιο, ύστερα από 300 χρόνια σκλαβιάς και 100 χρόνια apartheid, μπόρεσαν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες της ΗΠΑ. Μου παραχωρήθηκαν λοιπόν τα δικαιώματά του, αλλά το πιο σημαντικό ε, είναι ότι την ελευθερία μου την έδωσε το, η δυνατότητα να ασκήσω τα ε, καθήκοντά μου ως πολίτης και τις ευθύνες μου ως πολίτης. Από εκείνη τη στιγμή αποφάσισα να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να προσπίσω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το και όταν μου ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη και αρμοστία να καταστώ πρόσβυρα πρέσβυρα καλή λύσεω το 1986, θεώρησα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία να μετατρέψω σε πράξει τι πραγματικέ μου πεπιθήσει σε, ε, σε μια ευρύτερη κλίμακα. Και έτσι λοιπόν αγωνιστώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 30 χρόνια τώρα υψώνω τη φωνή μου ε, για να υπερασπιστώ τους πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Από την Νότια Αφρική στην Καμπότζη, το Ανατολικό Τιμόρ, τη Ρουάντα, την πρώην Γιουγκοσλαβία. Έχω συναντήσει τόσες χαροκαμένες μητέρες που χρειάστηκα ε, να, να θάψουν τα ίδια τους τα παιδιά. Πέρσι συνάντησα στην Ελλάδα μια μητέρα που ε, δακρύζοντας μου αφηγούνταν τη ζωή που εγκατέλειψε το μεγάλο ταξίδι στο οποίο αναγκάστηκε να καταφύγει. Το μόνο της μέλημα ήταν τα παιδιά της για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Πολλά παιδιά τη Συρία όμω έχουν χάσει πέντε σχολικέ χρονιέ λόγω τη τραγωδία αυτή. Πολλέ είναι οικογένειε που ακόμη έχουν μείνει στην Ελλάδα και περιμένουν η Ευρώπη να λάβει τελικά και γρήγορα μια απόφαση για την μετεγκατάσταση και να υλοποιήσει την απόφαση για την μετεγκατάσταση. Ο ύπατο αρμοστή Φίλιππο Γκράντι έχει πει ότι η αδυναμία τη Ευρώπη για υλοποίηση μια λογική απόφαση για την κρίση των προσφύγων οδήγησε στο χάο στα σύνορα και την κατάρρευση τη πίστη του κοινού των των πολιτών στη δυνατότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή. Δηλαδή, ουσιαστικά έδωσε δύναμη σε εκείνους που θέλουν να καταστήσουν τον πρόσφυγα από διοπομπαίο τράγο. Ε, το έγγραφο, το είπα της αρμοστίας, μια καλύτερη προστασία των προσφύγων, αποτελεί το πλαίσιο για ένα νέο όραμα για την διστράτευση της Ευρώπης και την προσήλωσή της για την αντιμετώπιση παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης. Όλες αυτές οι κρίσεις συνιστούν μεγάλες και φοβερές προκλήσεις. Πάνω απ' όλα όμως υποφέρουμε από μια ηθική κρίση. Φαίνεται σαν να κινούμαστε, να δρούμε, να αντιδρούμε χωρίς να έχουμε ηθικό μπούσουλα, χωρίς να έχουμε ένα όραμα, χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και γιατί. Έχουμε αφήσει να συνεχιστεί αυτό για πολύ καιρό. Έχουμε αφήσει τους εμπόρους του φόβου του μίσου, του αποκλεισμού να έχουν την ισχυρότερη φωνή και να προσδιορίσουν τι εθνικέ μα ταυτότητε. Οι λύσει που μα προτείνουν μπορεί να μα καλούν να κλείσουμε τα μάτια μα, να κλείσουμε τι καρδιέ μα, να κλείσουμε τα σύνορά μα στο κάθε τι και στον κάθε ένα που μπορεί να είναι διαφορετικό. Είχαν βοηθό βέβαια και συνένοχο και τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία είναι εθισμένα στην πρόκληση εντυπωσιασμού και κέρδου και που έχουν ξεχάσει εδώ και καιρό ότι καθήκον τους είναι να υπηρετούν τη δημοκρατία και να αποκαλύπτουν την αλήθεια. Αντί γι' αυτό ενθερίνουν την μείωση και την υποβίβαση του επίπεδου της, του πολιτικού διαλόγου. Εγώ πάντως είμαι πεπισμένη ότι οι κρίσεις αυτών των τόσο δύσκολων καιρών μας προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουμε τους ατομικούς μας φόβους και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κατά μέτωπο. Να κοιτάξουμε με θάρρος αυτούς τους ανθρώπους και τις καταστάσεις διαφορετικά και να δράσουμε διαφορετικά. Αυτές είναι οι εποχέ που ζούμε και πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Είναι καθήκον μας αυτό. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είχε πει ότι το τόξο της ιστορίας έχει μεγάλο μήκος Αλλά κλείνει προς τη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας και να ανακαλύψουμε και πάλι τις βασικές αξίες, τις αξίες πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί αυτή η Ένωση. Στο τέλος αυτής της μακράς και μαύρης νύχτας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Ευρώπη αναδύθηκε από τις τάχτες της Σαντοφίνικα. Δημιουργήθηκε μια νέα Ένωση. Δημιουργήθηκε για να φέρει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την επιμερία στους πολίτες της, καθώς και, το και για να προωθήσει την ισότιμη απόλαυση των αγαθών της ευημερίας, το δικαίωμα για ένα προστατευμένο περιβάλλον, σεβασμό των πολιτιστικών, θρησκευτικών και γλωσσικών διαφορών. Στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι η αδιέρετη και οικουμενική φύση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, οι αξίε τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δημοκρατία, αλληλεγγύη, ελευθερία και ισότητα τη ελευθερία δεν είναι δεδομένε και ότι πρέπει διαρκώ να επαγρυπνούμε. Το 1976 εγώ ακολούθησα την καρδιά μου και ένα νεαρό Σουηδό και μετακόμισα στην Ευρώπη. Πριν από 25 χρόνια περίπου αποφάσισα να γίνω πολίτη τη Ευρώπη για να έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το δύσκολο, περίπλοκο αλλά και τόσο υπέροχο εγχείρημα. Πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των συναυλιών μου έχω την εντύπωση ότι το κοινό και εγώ ε, ακούμε με ένα αυτή ότι δονούμαστε πάνω στην ίδια χορδή. Και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι η χορδή, η δόνηση πάνω στην οποία στηρίχθηκε και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Για μια μικρή σύντομη στιγμή θυμούμαστε ποιοι είμαστε. Ότι όλοι είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας και ότι είμαστε μέλη της οικογένειας της ανθρωπότητας. Πρέπει να είμαστε ατρόμητοι, να τολμήσουμε να κοιτάξουμε αυτόν, αυτόν που ονομάζουμε άλλον, και ας είναι απειλητικός και ας είναι διαφορετικός και να του πούμε αδελφή μου, αδελφέ μου, παιδί μου, Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατακτήσουμε το μίσος με περισσότερο μίσος. Και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, να χάσουμε την ανθρωπιά μας με το πρόσχημα ότι σώζουμε την ανθρωπιά μας ή την ανθρωπότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική στον κόσμο. Η μόνη ένωση κρατών που στηρίχθηκαν στην επιθυμία να μην επαναληφθούν ποτέ οι θηριωδίες του παρελθόντος. Και στόχο να οριστεί, στόχος να οριστεί η ειρήνη. Είμαστε μια μεγάλη ένωση, όχι γιατί είναι καλύτερε οι αξίες μας, αλλά γιατί οι αξίες μα είναι ανοιχτέ σε όλου και οικουμενικέ. Κλείσαμε τα 60, Όμω είμαστε ακόμη νέοι. Ο κόσμος τώρα μας χρειάζεται να αναλάβουμε την ηγετική θέση που μας ανήκει και που οφείλουμε να αναλάβουμε σε αυτή τη στιγμή. Στη χειρότερη στιγμή της κρίσης η καρδιά μου αισθανόταν συγκίνηση όταν έβλεπε τόσους πολλούς συμπολίτες μου Ευρωπαίους που έδειξαν τη συμπόνια, την αλληλεγγύη και την γενοδορία τους προς τις οικογένειες των προσφύγων. Μια δημοσκόπηση της ε, Διεθνούς Αμνηστίας το, 2016 απέδειξε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες φοβούνται λιγότερο τον πρόσφυγα από ότι τον φοβάται ο πολιτικός. Ως πρέσβυρα λοιπόν της ΥΠΑ της Αρμοστίας σας ζητώ να δείξετε την ίδια αλληλεγγύη με αυτή που θα θέλατε να δείξουν οι άλλοι στη δική σας την οικογένεια. Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω ένα προσφυγόπουλο στα μάτια χωρίς να δω το πρόσωπο των δικών μου παιδιών, των δικών μου εγγονιών. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε ε, όλες αυτές τις χώρες οι οποίες έξω από τα σύνορά μας ε, υποδέχονται με μεγάλη γενεοδορία κινήσεις και ροές προσφύγων. Όπως ο Λίβανος, χώρα 4 εκατομμυρίων που έχει υποδεχθεί 1,5 εκατομμύριο Σύρους και 500.000 Παλαιστινίους και πρέπει να δείξετε περισσότερη αλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και συμπόνια. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν σηκώσει τρομερό βάρο. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία έχουν μετεγκαταστήσει 70% των προσφύγων. Ω Ευρωπαία μητέρα και γιαγιά, σα καλώ να κάνετε το καθήκον σα. Να εκπροσωπήσετε τα παιδιά τη Ευρώπη και τι κοινέ μα αξίε. Στο θέατρο λέμε το θέαμα πρέπει να συνεχίζεται. Ε, ας πούμε ότι είναι η πρεμιέρα σήμερα ο αυτοανακηρυχθής πρωταγωνιστής της παγκόσμιας σκηνής μας είπε ότι είναι άρρωστος. Πρέπει λοιπόν να βγούμε στην παγκόσμια σκηνή και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι το σωστό. Ο καθένας από εμά έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, να παίξει. Είμαστε ενωμένοι και ισχυροί και μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Από την αδυναμία στη δύναμη, από την αδικία στη δικαιοσύνη, από το σκοτάδι στο φως, από την ειρήνη από τον πόλεμο στην ειρήνη, από το φόβο στην αγάπη μπορούμε να περάσουμε ενωμένοι. Δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη η εποχή και έχουμε υποχρέωση να επιτύχουμε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αποτύχουμε για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των παιδιών μας. Η αποτυχία είναι απαράδεκτη. Πρέπει να πλώσουμε το χέρι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect him to invite me. Βεβαίως. Δεν θα περιμένατε ότι με καλέσαν εδώ και δεν θα τραγουδούσα. Θα τραγουδήσω τώρα λοιπόν ένα πάνθισμα για τα προσφυγόπουλα μαζί με ένα πείμα του Western Shire, Σομαλού πρόσφυγα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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. Και τώρα με χαρά κατοσορίζω τον Ρόμπερτ Νενάσε, αυστριακό συγγραφέα που αφιέρωσε τη ζωή του στη συγγραφή για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμιοποίησης. Ο κ. Μενάσε είναι ο πραγματικός πρέσβης της Δημοκρατικής Χάρτας του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, μου υπόθηκε με τεπιμονής ότι πρέπει να μιλήσω 10 λεπτά. Είναι πολύ σύντομο σε σχέση με αυτά τα οποία πρέπει να σας πω. Αλλά 10 λεπτά από την άλλη πλευρά είναι και μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκεφτούμε ότι είναι 12 παρα 5. Διότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα βρίσκεται όντως στο χείλος της Αβίσου. Αλλά φαίνεται ότι έχουν σταματήσει τα ρολόγια. Διότι εδώ και χρόνια διαβάζω στις εφημερίδες ότι είναι 12 παρα 5. Οπότε, ακόμη και αν υπερβώ κατά πολύ το χρόνο μου, θα παραμείνει 10 ε, παρά 12. Business as usual δηλαδή, πολύ απλά. Διότι πέρα από όλες τις κοσμοϊστορικές αλλαγές πάντα υπήρχε business και αυτό είναι το usual, το σύνηθε. Όμως το ερώτημα είναι, εάν το business μετά μια καταστροφή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος συνοποίησης θα εγγυεί το ακόμη την ειρήνη με βάση τη δημοκρατία, την ισοτιμία και την κοινωνική ασφάλεια. Είτε εάν οι φίλοι θα γίνουν πάλι εχθροί και οι κυρίαρχοι πολίτες θα γίνουν πάλι αυταρχικά σύνολα που θα εμπλακούν σε μάχες για την κατανομή του εισοδήματος που μπορούν να οδηγήσουν σε εμφύλους πολέμους, σε εθνικούς πολέμους για τους ε, πόρους, ε, τα κεφάλαια, τις προσβάσεις στην αγορά και τις σφαίρες επιρροής. Δεν είναι πιθανό. Αν είμαστε ειλικρινείς ε, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ορισμένα φαίνονται ιδιαίτερα ζωφερά. Όμως Σήμερα θέλουμε να κάνουμε τέτοιες μαύρες σκέψεις και ανησυχίε για το μέλλον, όσο αιτιολογημένες και αν είναι. Τώρα εορτάζουμε μια επέτειο, την 60η επέτειο τη υπογραφή των συνθηκών της Ρώμης. Επέτη σημαίνει εορτές. Σε επίσημες εκδηλώσεις όπου περήφανοι ε, δεν είναι τώρα η ώρα για ε, απειλές, αλλά πρέπει να πούμε ε, κοινό το παλόγια χαράς. Όμως ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ καλοί και βάσιμοι λόγοι για υπερηφάνεια και ικανοποίηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όποιο ε, θυμάται την υπογραφή των ε, συνδικών τη Ρώμη, όποιο θυμάται τι επέτυχαν οι ιδρυτέ, τι προθέσει, ε, τι απόψει του, όποιο τι εορτάζει, μέσω του εορτασμού διατυπώνει έντονη κριτική στη σημερινή κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν θυμηθούμε τι συνθήκε τη Ρώμη, γίνεται επώδυνα σαφέ ποια είναι η θέση των σημερινών Ευρωπαίων πολιτικών τι ξέχασαν ή ποτέ δεν κατάλαβαν δηλαδή. όποιο υμνεί του ιδρυτές στην ουσία υποβάλλει τους κληρονόμους τους σε ισοπεδωτική κριτική. Σκεφτείτε το εξή. Αν ερωτήσετε του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ή του υπουργού των ε, κρατών μελών τη Ένωση που σήμερα λαμβάνουν αποφάσει στο Συμβούλιο, ποιε ήταν οι ιδέε και προθέσει των πολιτικών που υπέγραψαν τι συνθήκε τη Ρώμης θα διαπιστώσετε δεν τις γνωρίζουν. Και αν ε, τους τις πούμε, τότε απαντάνε, μα τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Αυτές είναι τρέλες, ε, παλαβομάρες, ε, ουτοπικές. Ναι, αυτό λένε οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι σήμερα στα Ινία και γι' αυτό θεωρούν ότι είναι ρεαλιστές. <clears throat> Γιατί δεν έχουν όραμα για το μέλλον, απλώς διαχειρίζονται κρίσεις, τις οποίες αυτοί τόσο ρεαλιστικά προκάλεσαν οι ιδρυτές με βάση την ιστορική εμπειρία προσπάθησαν να δουν μακριά στο μέλλον αλλά σήμερα στην ουσία ξεχνάμε και προσπαθούμε να επιμηκύνουμε τη σημερινή κακή κατάσταση. Αυτή είναι η ουσία της κρίσης. Και γι' αυτό είναι τώρα 12 παρα 5. Γιατί ήταν παλαβή η Ποια ήταν η τρελή ουτοπία. Έχω μόνο 10 λεπτά. Τώρα μου έχουν μείνει 8. Και σε αυτά θα σα πω μόνο τα απολύτω απαραίτητα. Αν και ίσω να μην είναι πολύ εορταστικά. Θέλω δύο λεπτά πρώτα απ' όλα να σα υπενθυμίσω τι θα έπρεπε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το πιστοποιητικό γέννησή τη, <clears throat> που είναι οι συνθήκε τη Ρώμη. Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, ο ευρωπαϊκό εθνικισμό οδήγησε σε ισοπεδωτικούς, δύο ισοπεδωτικού παγκόσμιου πολέμου, και στα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα μέχρι και το ίδιο το Auschwitz. Ο ευρωπαϊκό ε, πολιτισμό είχε καταστραφεί. Από αυτήν την εμπειρία έπρεπε να εξαχθούν διδάγματα. Δεν έπρεπε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μόνο αυτή η φράση. Αυτό το ποτέ πια ήταν μια υπόσχεση που θα έπρεπε να ισχύει αιώνια. Το ερώτημα είναι πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Αυτά τα εχθρικά μεταξύ τους ε, έθνη να συμφιλειωθούν και να υπερβούμε τον εθνικισμό τους ώστε να υπάρχει μόνιμη ειρήνη και ελεύθερη συμβίωση σε αυτήν την έρημο που την, την Ήπειρο που την είχε ερημώσει η ιστορία. Οι ιδρυτές της ΕΕ είχαν διαπιστώσει ότι οι συνθήκες ειρήνης και οι συνασπισμοί εθνικών κρατών δεν εμπόδιζαν τους πολέμους. Οπότε προέκυψε η ιδέα ότι πρέπει να υπάρξουν στενές και σύνθετες σχέσεις μεταξύ των οικονομιών των εθνικών κρατών, ώστε να υπάρχει ένα σύστημα αλληλεξάρτησης που τελικά να οδηγήσει σε μια συνεργασία στη βάση αναγκαίων κοινών συμφερόντων. Ούτως ώστε οι εθνικοί απομονωτισμοί που ιστορικά είχαν αποδειχθεί λανθασμένοι και επικίνδυνοι να καταστούν αδύνατοι. Ωραία. Γνωστή αυτή η ιστορία. Αυτός είναι όμως και ο λόγος γιατί οι πολιτικοί θύνοντες και από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι πολίτες στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς μια καλύτερη οικονομική κοινότητα ότι ο πυρήνα τη είναι μια κοινή αγορά. Την οποία όμω παρανοούν. Γιατί νομίζουν ότι είναι απλώ πλεονέκτημα για τι εθνικέ του οικονομίε και για τα εμπορικά του ισοζύγια. Αλλά την πολιτική ένωση τη βλέπουν με όλο και περισσότερη δυσπιστία, ότι θα του αφαιρέσει δικαιώματα, ότι θα καθορίζουν άλλη τη μοίρα του, ότι θα απειλήσουν τη λεγόμενη εθνική κυριαρχία. Γι' αυτό τα εθνικά συμφέροντα τα υπερασπίζονται ακόμη και σε αυτή την υποτίθεται κοινή αγορά. Για παράδειγμα, υπερασπίζονται τις εθνικές αγορές εργασίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες και οι εκπρόσωποι τους πέφτουν και πάλι στην παγίδα του εθνικισμού, που υποτίθεται ότι έπρεπε να τον υπερβούμε. Οι ιδρυτές, όμως, πριν από 60 χρόνια, είχαν την πρωτοπόρο άποψη ότι ο εθνικισμός πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του. Δηλαδή, πρέπει, στη τελευταία ανάλυση, να υπάρξει σταδιακή υπέρβαση των εθνικών κρατών αυτή η άποψη είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα και να θυμηθούμε. Η διασφάλιση ειρήνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη βάση ένα εγχείρημα για την υπέρβαση των εθνικών κρατών. Ωραίο να λέμε εξασφάλιση της ειρήνης. Και μπορεί πολλοί να το θεωρούν ε, και ανιαρό. Αλλά δεν είναι καθόλου ανιαρό. Γιατί έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι αντιφάσεις που περιγράφουμε σήμερα ως κρίσεις είναι κατανοητές μόνο να σκεφτούμε ότι στην αρχή υπήρχε η συγκεκριμένη ουτοπία ή διαδηλωμένη πρόθεση να επιτευχθεί διαρκής ειρήνης μέσω της υπέρβασης των εθνικών κρατών. Έξι λεπτά μου μένουν ακόμα. Οι συνθήκε τη Ρώμη είναι το πιστοποιητικό γέννηση της Ευρωπαϊκή Ένωση που έπρεπε λοιπόν να είναι ένα εγχείρημα για την υπέρβαση των εθνικών κρατών. Πρέπει να το πω επανειλημμένα αυτό. Γιατί αυτό ακριβώ είναι που έχουν ξεχάσει σήμερα οι ηθήνοντε στην Ευρώπη. Ή απλώ δειλά το αποσιωπούν οι συνθήκε τη Ρώμη. Σημαίνουν λοιπόν πιστοποιητικό γέννηση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το οποίο κοινοβούλιο στην αρχή δεν είχε καθόλου δικαιώματα και αρμοδιότητε. Κι όμω ήταν το πιστοποιητικό γέννηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια πολιτική επανάσταση επανάσταση, συγγνώμη. Διότι έτσι προέκυψε το πρώτο άμεσα εκλεγμένο υπερεθνικό κοινοβούλιο. Και τι έννοια μπορεί να έχει ένα υπερεθνικό κοινοβούλιο, αν όχι αυτή, ότι η προοπτική του είναι να υποκαταστήσει τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το χειροκροτήσετε ε, όταν υπενθυμίζω αυτή την ιδέα. Ο την, ε, η αυτοβιογραφία του Σαστή Συστήνο, στα απομνονέματα του, εκεί που αναφέρεται στη διαπραγματεύση για τη συνθήκη τη Ρώμη, είπε και παραθέτω, υπήρχαν πολλέ εθνικέ αντιστάσει. Αλλά τελικά είχαμε και την πείρα ότι τα έθνη και οι πολιτικοί τους θεσμοί είχαν αποδείξει αποφασιστικά ότι δεν είναι επαρκής για να επιτευχθεί η ειρήνη και το κράτος δικαίου σε μόνιμη βάση. Οπότε εξαγάγαμε από αυτό όλα τα άλλα συμπεράσματα. Να επιτύχουμε το πολιτικά αμέσως εφικτό και κατόπιν σταδιακά να ε, δημιουργήσουμε και άλλα πολιτικώς εφικτά. Κλείνω την παράθεση. Και ο Βάλτερ Χάλσταϊν, ένας από τους ε, πνευματικούς πατέρες των ε, συνδικών της Ρώμης, είπε στον περίφημο λόγο του στη Ρώμη και πάλι παραθέτω ότι αποφασίζουν αυτά τα νεοεδρυθέντα ευρωπαϊκά όργανα και επιχειρούν να εφαρμόσουν έχει ως στόχο να οργανωθεί μία μεταεθνική Ευρώπη. Πόσο μεγάλη είναι η σημερινή κρίση, η αντίδραση σε αυτό. Μπορούμε να το μετρήσουμε με αυτούς τους στόχους. Μπορείτε να σκεφτείτε έναν από τους ε, κυρίους γερμανικούς ηθήνοντες. Έναν ή ένα και μόνο. Να σκεφτείτε που θα μπορούσε, θα τολμούσε σήμερα να πει αυτή τη φράση του Βάλτερ Χάλσταϊν, του Γερμανού Βάλτερ Χάλσταϊν. Μπορείτε να σκεφτείτε κανέναν αρχηγό κρατών και κυβερνήσεων στην Ευρώπη που θα συμφωνούσε με αυτή την πρόταση. Βλέπετε. Θα μας έλεγαν ότι είμαστε τρελοί, ότι είναι πάλα όλα αυτά. Οι πολιτικοί θύνοντες που σήμερα φέρουν την ευθύνη για την ευρωπαϊκή πολιτική, έτσι λοιπόν είτε ξέχασαν είτε ποτέ δεν κατάλαβαν την ευρωπαϊκή ιδέα. Γιατί, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί δεν λένε περί πρόκειται, γιατί κάνουν αυτού του πανηγυριώτικου λόγου όπου λένε ότι χρειάζεται η Ευρώπη αλλά δεν εξηγούν τι είναι η Ευρώπη. Γιατί ε, μιλάνε για τι ευρωπαϊκέ αξίε και για την ειρήνη και επιχειρούν να το επιβάλλουν μέσω περιορισμού των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω καταστάσεων έκτακτη ανάγκη, μέσω τη συμμετοχή σε πολέμου άλλων. Γιατί θέλουν οι, οι να είναι γελιοποίηση του εαυτού της αντί να, την, προσπαθούν να την εφαρμόσουν. Γιατί δεν προσπαθούν να υπάρξει ένα μεταεθνικό σύνταγμα, να επεκταθεί περισσότερο, να προωθηθεί περισσότερο η μεταεθνική δημοκρατία προς ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος. Γιατί κρυβόμαστε στην αμηχανία μας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κρυβόμαστε κυρίως πίσω από εθνικές σημαίες και τραγουδάμε εθνικούς ύμνους κρατικού αντί να προωθούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Γιατί πάντα με φαινομενική πικρία λέμε ότι η Ευρώπη δυστυχώς δεν είναι να εξηγηθεί στους πολίτες. Γιατί δεν υπάρχει καμία αφήγηση, κανένα αφήγημα. Γιατί να μην μπούμε δυνατά. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε ένα αφήγημα. Έχουμε. Άνθρωποι όπως ο Ζάμο Νέο, ο Βάτερ και ο Ζάκ Δελόρ το διατύπωσαν. Απλώς ε, στην καθημερινή πολιτική ξεχάσαμε να τα λέμε αυτά την ιδέα ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι η υπέρβαση των εθνικισμών. Στο τέλος η υπέρβαση των εθνών. Τι είναι τόσο περίπλοκο και ακατανόητο σε αυτό. Γιατί να μην το πούμε δυνατά. Δεν είναι θέμα της ε, κυριαρχίας των Ευρωπαίων πολιτών ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι μάλλον το θέμα και όχι η ε, κυριαρχία των κρατών. Γιατί δεν το λέμε αυτό με αυτοπεποίθηση. Γιατί με αμηχανία κοιτάμε όταν κερδίζουν ε, επιρροή οι εθνικιστές κάθε είδους. Γιατί κάνουμε παραχωρήσεις αντί να τους αντιμετωπίσουμε με τα καλύτερα επιχειρήματα. Εμείς έχουμε την ιστορική γνώση του τι έκανε ο εθνικισμός. Κατέστρεψε τον, ε, την Ήπειρό μας και προκάλεσε ανίποτα δεινά για ε, αμέτρητα εκατομμύρια συμπολιτών μας. Ο εθνικισμός δεν είναι όμορφη ουτοπία. Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι ιστορικό έγκλημα. Αλλά η μεταεθνική εξέλιξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο στα μικρά βήματα που έχει επιτύχει μέχρι ώρα έφερε ειρήνη και ευημερία στην Ήπειρό μα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι που βάλτωσε σε αυτέ τι αντιφάσει. Το ότι τα κράτη-μέλη δηλαδή ξεκίνησαν πάλι να προσπαθούν να, ε, ε, να προωθήσουν τα εθνικά τους ε, ε δικαιώματα κυριαρχίας κατά της Ευρώπης. Όλες οι κρίσεις στην Ευρώπη είναι σήμερα προϊόν αυτής της αντίφασης. Ο εθνικισμός δεν είναι η λύση, είναι το πρόβλημα. Ο Στέφαν Τσβάικ έγραψε το 1913 τα εξή. Είτε θα συντρίψουμε τον εθνικισμό, είτε θα καταστραφεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ξέρουμε τι συγκρούσεις προέκυψαν μετά. Οι ιδρυτές ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματο ε, από την πείρα με τον εθνικισμό μετά το δεύτερο πόλεμο μεταξύ του 1914 του 1945 εξήγαγαν τα σωστά διδάγματα. Και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά στους συμπολίτε μας. Η ιστορική πείρα που έχουμε δικαιολογούν τους σημερινούς συμβασμούς με τους εθνικισμούς στα κράτη-μέλη. Φυσικά όχι. Αντίθετα. Έχουμε ικανούς ε, υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ε, αγωνιστικούς ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή γνώμη που να στηρίζει την καταπολέμηση της επανεθνικοποίησης της Ευρώπης. Αυτοί που θέλουν να ε, μας ξαναγυρίσουν πίσω μας φέρνουν τον πόλεμο. Ο συμβασμός μαζί τους θα μας φέρει μία μακρά και επώδυνη παρακμή. Η αναζωγόνηση της ευρωπαϊκής Ουτοπία είναι η λύση. Είμαστε τώρα 60 χρονών και ήδη έχει κάνει πολλά και αποδείχθηκε ότι είναι συγκεκριμένη και ρεαλιστική ουτοπία. Και η ιδέα της ε, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τις ιδέες αυτών που θεωρούν σήμερα ότι είναι πραγματιστές. Τώρα μου μένουν τρία λεπτά. Ξέρω ότι και στο σώμα αυτό υπάρχουν ε, ευρωβουλευτέ που δεν αισθάνονται ότι είναι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποι των εθνών τους. Επιδιώκουν να παρεμποδίσουν την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αλλά δεν θα μπορέσουν τελικά να τη σταματήσουν. Και ξέρω φυσικά επίσης ότι πολλοί πολίτες στην Ευρώπη ποθούν την αποκατάσταση της ε, κυριαρχία των εθνικών κρατών. Οι Ευρωπαίοι όμω μεταξύ μα δεν θα πρέπει να εξαπατηθούν από αυτά. Στον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, Κρίσει, απειλέ, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι πρωτοφανή και δεν τα καταλαβαίνουμε ακόμη. Και πολλοί πιστεύουν ότι το εθνικό κράτος ε, είναι σαν ε, ένα σπίτι και ότι αυτοί είναι οι νοικοκύριδε. Και θέλουν ακριβώ αυτό να είναι. Νοικοκύριδε στο σπίτι του, Ακόμη και αν ζουν στο υπόγειο. Ακόμη αν είναι στο δωμάτιο υπηρεσία και ποτέ δεν πρόκειται να ανέβουν στου πάνω ρόφου, πάντα με περισσότερη αποφασιστικότητα, με περισσότερη πικρία θέλουν να εκπροσωπηθεί η πολιτική τους. Ότι είναι νοικοκύριδες. Και θεωρούν, θεωρούν πραγματικά ότι είναι κύριοι της ιστορίας τους και δεν είναι πλέον θύματα. Όποιος ενισχύει αυτούς τους προφόρους, συγγνώμη, όποιος προσπαθεί να πάρει τις ψήφους αυτών, κάνει για άλλη μια φορά σοβαρό λάθος. Διότι η μεταεθνική εξέλιξη θα γίνει, είτε το θέλουν είτε όχι και δεν ασχολείται με νοικοκυριά. Η κυριαρχία των εθνικών κρατών αντικειμενικά καταργείται. Το πολιτικό περιθώριο λιγμών των εθνικών κυβερνήσεων μειώνεται. Τα εθνικά σύνορα εξαφανίζονται. Ακόμη και αν κάποιε κυβερνήσει προσπαθούν να τα αποκαταστήσουν. Η ιδέα ότι το έθνος είναι μια κοινότητα ισοτήμων γίνεται ε, στην πράξη σήμερα αυτό που θεωρητικά πάντα ήταν. Καθαρός μύθος. Όλα τα φαινόμενα που σήμερα καθορίζουν τη ζωή μας ή μας πιέζουν είναι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διεθνικά. Οι αλυσίδε παραγωγή, οι αλυσίδε τροφίμων, οι χρηματοδοτικέ ροέ, τα οικολογικά προβλήματα, το ίντερνετ, η μας πιεζουν ειναι εδω και μεγαλο χρονικο διαστημα διεθνικα οι αλυσιδε παραγωγη οι αλυσιδε τροφιμων οι χρηματοδοτικε ρομε τα οικολογικα προβληματα το ιντερνετ η παρακολουθηση και οι απειλέ κατά των δικαιωμάτων, η τρομοκρατία, ό,τι και αν είναι. Όλα αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν σταματάνε στα εθνικά σύνορα και δεν μπορούν εντό εθνικών συνόρων να επιληθούν. Όλα όσα εμπλουτίζουν τη ζωή μας και την κάνουν αξιόλογη. Η τέχνη, ο πολιτισμός, η επιστήμη, η ανταλλαγή ιδεών και καινοτομία. δεν σταματάνε σε εθνικά σύνορα. Τα εθνικά σύνορα δεν ε, προστατεύουν την, ε, τον πολιτισμό και το πνεύμα, αντίθετα τα καταπνίγουν. Αυτά πρέπει να πούμε σε αυτούς που αφιβάλλουν, στους σκεπτικιστές, σε όλους που ε, πάνε στους εθνικιστές. Αυτά πρέπει να τους πούμε. Η μεταεθνική μετάβαση μπορεί να τη σταματήσει κανεί βία για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Ρωτήστε τους πολίτες ξεκάθαρα, θέλετε να σταματήσετε την εξέλιξη και να πληρώσετε ως αντίτυπο την ανέχεια των περισσότερων είτε θέλετε αυτή την εξέλιξη μόνο απρόθυμα και με λάθος συμβασμούς να την ε, βαλτώσετε σε μόνιμες κρίσεις είτε θέλουμε να διαμορφώσουμε εμείς με τον σωστό τρόπο αυτή την εξέλιξη και φυσικά όλοι θέλουν, ο οποίος έχει σώαστας φρένας να διαμορφώσει τις συνθήκες της ζωής του, όχι να τις υφίσταται αυτό είναι σαφές από κοινού θα παρεύουμε στις διεθνικέ διαδικασίες μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια διεθνική πολιτική μία ενωσιακή πολιτική, μία ευρωπαϊκή πολιτική στο πνεύμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 60 χρόνια επέτυχε αξιόλογες νίκες ε, στην καταπολέμηση, στη μάχη για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινοβουλευτισμού, ούτως ώστε να επιτύχουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ναι, αυτό βεβαίως θέλουμε και πρέπει να το γιορτάσουμε. Αλλά πολύ χρόνο για γιορτές ε, και για την ειδονή της επανάπαυσης δεν έχουμε. Μετά από 60 χρόνια τώρα έχω 10 λεπτά για αυτό το λόγο. Άρα σωστό είναι ε, να σας κάνω έκκληση ότι και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο για να παρεμποδίσετε να αποτύχει αυτό που σήμερα εορτάζουμε. Στα τελευταία λοιπόν λεπτά που έχω στη διάθεσή μου τώρα που είναι 12 παρά ένα λεπτό, πολύ σύντομα να συνοψίσω αυτά που ελπίζω και αυτά που φοβάμαι. Πολλά από αυτά που οι ιδρυτές θεώρησαν απαραίτητα και που κατέγραψαν στις συνθήκες δεν ήταν δυνατά να υλοποιηθούν τότε. Η Δημοσιονομική Ένωση, η εναρμόνιση των κοινωνικών παροχών, μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, η ανάπτυξη μιας κοινότητας της άμυνας κτλ. Όλα αυτά λοιπόν έμειναν πόθη τότε. Έμειναν ένα πρόσθετο πρωτόκολλο. Σήμερα είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να υλοποιηθούν. Και να και σε εσά κύριε και κύριοι βουλευτές αυτήν τη μεγάλη προοπτική να την ενσωματώσετε, να μην τη λησμονήσετε στην καθημερινή σας δουλειά, στη δουλειά της ρουτίνας. Αντιθέτως να την οργανώσετε με την πολιτική πίεση και να την υλοποιήσετε επιτέλους και να πόκειτε σε όλους εσάς τα μέλη της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ξεπεράσετε τα δημοκρατικά ε, ελλείμματα της Ένωσής μας, να εξαλείψετε τις αφόρητες αντιφάσεις της που αποτελούν και την αδυναμία δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε την ιδέα μιας μεταεθνικής Ευρωπαϊκής Εθνοσυνέλευσης, αλλά εκλέγουμε με βάση μια εθνική εκλογική λίστα. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει ως υπερεθνικός οργανισμός, ως υπερεθνικό όργανο το καθήκον της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά η ηγεσία της ορίζεται από, τα, από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες Θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι πολίτε και πρέπει να είμαστε. Αλλά δεν έχουμε, ανάλογα με το κράτο μέλο στο οποίο γεννιόμαστε, τα ίδια δικαιώματα, τι ίδιε ευκαιρίε ζωή, την ίδια στάθμιση ακόμα και ειδικό βάρο στη ψήφο μα. Ω Ευρωπαίοι πολίτε, λοιπόν, έχουμε ακόμη εθνικό διαβατήριο. Εάν οι Βρετανοί είχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια, θα μπορούσε βέβαια η Βρετανική κυβέρνηση να αποφασίσει να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Αλλά οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον δεν παραδώσουν τα διαβατήριά του, θα παρέμεναν πολίτε. Γιατί είναι ε, πολίτε τη Ευρώπη. Γιατί είναι Ευρωπαίοι. Όλα αυτά είναι αφόρητες αντιφάσεις και, προξενούν αντιπαραγωγικές κρίσεις οι οποίες ε, στερούν την εμπιστοσύνη του πολίτη στη λογική βάση της Ένωσης και το εγχείρημα της ε, ενοποίησης. Πρέπει να αρθούν λοιπόν αυτές οι αντιφάσεις, πρέπει να μετεξελιχθεί η Ένωση και αυτό είναι λεπτομέρεια κυρίες και κύριοι σε σχέση με το επίτευγμα εκείνων την εποχή των συνθήκων της Ρώμης που μπόρεσαν αντιμέτωποι με το πνεύμα των καιρών να ξεπεράσουν τη δυσπιστία του ε, νικητή έναντι του ηττημένου, να ξεπεράσουν την ανάγκη του θύματος για ρεβανσισμό. Και θέλω να το καταστήσω πολύ το σαφές. Όσο δύσκολο και αν το καθήκον αυτό το σημερινό το δικό σας, είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα καθήκοντα που επιτέλεσαν οι ιδρυτές. Αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ πιο κατεπίγουσα και οξία η ανάγκη να υλοποιήσετε αυτό το καθήκον για να μην οδηγηθούμε στην καταστροφή. Γιατί πεθαίνουν ένας-ένας ε, οι επιζήσαντες της ευρωπαϊκής αυτής καταστροφής που θα μπορούσαν με την προσωπική τους μαρτυρία να εξηγήσουν πόσο απαραίτητο είναι να αγωνιστούμε κατά του εθνικισμού. Να δώσουμε την υπόσχεση λοιπόν που δόθηκε πριν από 60 χρόνια ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ το ποτέ πια να γίνει μόνο λόγια κενά και ότι θα υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση για να προχωρήσουμε στο μέλλον της εποχής μας αυτό που διαμορφώθηκε μέσα από ένα ιστορικό δίδαγμα, μια ιστορική διαδαχή. Χωρί ημερομηνία λήξεω. Και να αποχτύπησαν τα 10 λεπτά. Σε ιστορικέ διαστάσει, πολύ λιγότερο από το ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου ο χρόνο που δόθηκε για την αξιολόγηση των 60 ετών. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου, ξεπερνώντα το χρόνο ομιλία μου, με τα τελευταία λόγια, να εκφράσω το φόβο μου. Το φόβο μου ότι στο εγγύ μέλλον ο λεγόμενο πολιτικό πραγματισμό θα προδώσει την πολιτική ιδέα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και θα τη βλάψει αμετάκλητα. Φοβούμε ότι παραδείγματι εσείς θα συμβάλλετε στην εγκατάλειψη, στην προδοσία των ε, Σκοτσέζων που θέλουν να είναι Ευρωπαίοι για να ικανοποιήσετε τους εθνικιστές του Λονδίνου. Και έτσι θα ενισχύσετε τις φυγόκεντρες δυνάμεις που θέτουν σε κίνδυνο το έργο της ενοποίησης της Ευρώπης. Ένα παράδειγμα μόνο των φόβων μου, ότι και των μελημάτων μου ότι η ιδέα των ιδρυτών της Ευρώπης έχει λησμονηθεί. Η ιδέα έλεγε ότι πρέπει τα εθνικά κράτη να εκλείψουν και θα εκλείψουν για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο των ελεύθερων περιφερειών με ένα νομικό καθεστώς που θα έχει μια κοινή ένωμη τάξη ε, πεφωτισμένη ε, η οποία στην μετεθνική Ευρώπη θα αποτελεί το θεμέλιο μιας ειρηνική, ενός μέλλοντος ειρηνικού και ευημερούντος. Και παραπέμπω και πάλι στα λόγια του Βάλτερ Χαλστάιν δεν πρέπει να περιοριστούμε στην εξάλληψη των παραδεγμένων συνόρων για να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων. Πρέπει πέραν αυτού να αντισταθμίσουμε τις παραδοσιακές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και να διορθώσουμε και όποιες νέες ανισότητες προκύψουν πάλι θα είμαστε σε αντίφαση, σε αντίφαση με τους στόχους των συνθήκων της Ρώμης που ήταν η μείωση της οικονομικής απόστασης μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και ταυτόχρονα η προστασία των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Η πολιτική λοιπόν υπευθυνότητα, η περιφερειακή πολιτική υπευθυνότητα της κοινότητας ισχύει όχι μόνο για τους χώρους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στον κίνδυνο της ε, υπερεξέλιξης αλλά πάνω απ' όλα στους χώρους που είναι πιο αδύναμοι οικονομικά. Η οικονομική και η κοινωνική πολιτική λοιπόν πρέπει να είναι στο επίκεντρο μιας περιφερειακής πολιτικής, μιας περιφερειακής πολιτικής που πρέπει να ε, διαπερνά όλες τις πολιτικές εγκάρσεις, αλλά ταυτόχρονα και αντίστροφα μια περιφερειακή πολιτική πρέπει να είναι εκείνη η οποία θα υλοποιεί την ολοκλήρωση τη της ευρωπαϊκής κοινωνικής και ε, οικονομικής πολιτικής. Μια ένωση λοιπόν για την ειρήνη μπορεί να υλοποιηθεί τώρα, μια ένωση η οποία μπορεί να είναι αδιανόητη αυτή τη στιγμή με ε, μέσα στην περίοδο που θεωρούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ε, κινδυνεύσουν τα κράτη να βρεθούν αντιμέτωπα στρατιωτικά το ένα με το άλλο. Όμως, όμως μια ένωση για την ειρήνη μόνο κατόνομα μπορεί να είναι τέτοια εάν δεν εξασφαλίζει και την κοινωνική ειρήνη στην Ήπειρο αυτή. Μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα το οποίο θα εξασφαλίζει ελευθερία, ισοδικία και ισότιμη πολιτική συμμετοχή για κάθε Ευρωπαίο πολίτη, για κάθε Ευρωπαία πολίτη, ανεξαρτήτως της, ε, του Εθνικού Διαβατηρίου που φέρει. Και αυτό είναι στο επίκεντρο του καθήκοντος για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ρεσπούμπλικα, μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το συναρπαστικό καθήκον που έχετε εσείς, επομιστεί κυρίες και κύριοι. Η Ευρώπη να καταστεί μια παγκόσμια πολιτική avant-garde. Να πανηγυρίσετε, να πανηγυρίσετε όμως. Οι πανηγερικές εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα. Και σε 10 χρόνια που θα έχουμε να εορτάσουμε τα 70 χρόνια από τις συνθήκες της Ρώμης, θα εορτάσουμε τα μεγάλα βήματα που θα έχουμε εντωμεταξύ υλοποίηση. Τι λείπει. Λείπει ακόμη αυτό που θα το προσθέσω, μια φράση γεμάτη αγωνία. Ζήτω και επιτρέψτε μου με μία λέξη να πω ζήτω η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και επιτρέψτε μου ακόμη να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι είναι ουσιοδέστατοι για τη λειτουργία αυτής της Ένωσης. Θα είμαι πολύ σύντομος για τα συμπεράσματα και την κατάληξη αυτής της εκδήλωσης. Συμπερασματικά, κλείνοντας αυτό το πρώτο μισό μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στα 60 χρόνια ιστορία των συνθήκων, και πρέπει να προσθέσουμε και τα 10 για την προετοιμασία τους, θα έπρεπε να πω και κάποια πράγματα για το μέλλον της Ευρώπης, που είναι το λίκνο του πολιτισμού. Η ιστορία μας είναι πάνω απ' όλα μια ιστορία δέσμευση για την ελευθερία. Για αυτή την ελευθερία πέθαναν εκατομμύρια Ευρωπαίων, αλλά και εκατοντάδε. χιλιάδες Αμερικανοί, Καναδοί και Αυστραλοί στρατιώτε. Και προ αυτού εκφράζουμε την αμέριστη ευγνωμοσύνη μα για την ελευθερία, χάρη στην οποία αποκτά δουλειά, Χτίζει το μέλλον σου, την ευημερία σου, την οικονομία, τα σπίτια, τι υποδομέ. που αποκτήσαμε ξανά και χάρη στο σχέδιο Μάρσαλ. Είναι η ελευθερία που είναι η βάση του μεγάλου οικονομικού μα χώρου, όπου εμπορεύματα, κεφάλαια, υπηρεσίε και κυρίω εργαζόμενοι και άτομα μπορούν να κινηθούν χωρί σύνορα. Ακριβώ 60 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η μεγάλη μα περιπέτεια. Δεν ήταν εύκολο Πολλές φορές σταματήσαμε απογοητευμένοι προς τα σε κρίσεις. Όμως, ποτέ δεν, καταλ... δεν καταλήψαμε την προσπάθεια, δεν αποθαρρυνθήκαμε, ξεπεράσαμε τις δυσκολίες, τη πιστία την έλλειψη κατανόησης. Χτίσαμε πάνω στην εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Μαζί δουλέψαμε για πιο ανοιχτό, ένα πιο ανοιχτό κόσμο, με περισσότερα δικαιώματα, βοηθώντας για να βγουν από το σκοτάδι της δικτατορίας τόσες χώρες της Υπήρου μας. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την ελευθερία και για την πραγματική μας Ευρώπη που δημιούργησε ευημερία, θέσεις απασχόλησης, που κατέστησε το μεταξύ μας πόλεμο εφιάλτη του παρελθόντος. Αυτός ο μεγάλος χώρος συναντήσεων, ανταλλαγών, έχει βαθιές ρίζες. Είναι η ιστορία μας. Εμείς είμαστε οι έμποροι της Κρήτης, της ε, Καρχιδόνας, είμαστε οι φιλόσοφοι, οι γλύπτες, οι μαθηματικοί της Αθήνας, του Κρότονα, των Σιρακουσών, οι νομικοί και οι μηχανικοί της Ρώμης. Ο πολιτισμό μα γεννήθηκε στι ακτέ τη θάλασσα, στα νησιά, στι όχθε των ποταμών. Πλουτίσαμε χάρη στην ανταλλαγή, στη διαλεκτική, τη συνεχή, που είναι φυτόριο των ιδεών, ανταλλαγή σκέψεων, χάρη στι τέχνε και στι ε, επιστήμες. Μεταλαμπαδεύσαμε την αρχαία γνώση τόσων ταγμάτων ξεκινώντα από του ε, Βενεδικτίνου. Γεννήθηκαν έτσι τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ζωγόνο δύναμη ενό νέου ουμανισμού. Η αναγέννησή μα μα ενέπνευσε αυτέ τι γνώσει. Βγήκαμε έξω και γίναμε Βενετσιάνοι, Φλαμανδοί, έμποροι, Τοσκάνοι, τραπεζίτε. Μεγάλοι με που επένδυσαν στην τέχνη, στον πολιτισμό, προσελκύοντα και προσκυνητέ. Αυτό ο μεγάλο ευρωπαϊκό χώρο προσέλκυσε μεγάλου καλλιτέχνε, λόγιου, φιλόσοφου, μουσικού, Επιστήμονε που η μένα έμαθαν του δε. Ενέπνευσαν και εμπνεύστηκαν. Ο Καραβάτζου και ο Ρέμπραντ, όπω ο Βιβάλτη και ο Μπαχ, ο Σέξπιρ και ο Μολιέρο είναι ενωμένοι από έναν ακατάλληλο δεσμό, όπω ο δάντη, που είναι και ο Θερβάντες που είναι ανήκει όχι μόνο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό ο χώρο υπάρχει ακόμα. Ε, και υπάρχει πάντα μια νέα ευκαιρία. Είναι η Ευρώπη που πρέπει να ανοίξουμε στου νέου. θα πρέπει να τους δωρήσουμε τη δυνατότητα να μην εγκαταλείψουν τα όνειρά τους. Θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να πιστέψουν στο μέλλον. Θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να βρουν δουλειά. Γιατί χωρίς δουλειά δεν υπάρχει αξιοπρέπεια και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα παιδιά μας να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Γιατί είπα και πριν ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η ιστορική αγορά, δεν είναι μόνο το ευρώ. Δεν είναι μόνο το τραπεζικό σύστημα, δεν είναι μόνο η οικονομία. Η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο από αυτά. Πριν γίνει Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο πρώτος Ισπανός ε, αυτοκράτορας, ο Τραϊανός, ζήτησε από τον πατέρα του Μπορεί ένας Ισπανός να γίνει Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ο πατέρας του το απάντησε. Η Ρώμη δεν είναι μια πόλη. Η Ρώμη είναι ένα μοντέλο πολιτισμού. Και ήταν τότε. Σήμερα, εάν τα παιδιά μας μας ρωτήσουν «Μπαμπά, μαμά, η Ευρώπη είναι οι είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Είναι η πολιτική. Είναι οι τράπεζες. Εμείς έχουμε το καθήκον νομίζω να απαντήσουμε στα παιδιά μας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, όχι. Η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ιδανικό. Η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός μας. Η Ευρώπη είναι η ταυτότητά μας. Η Ευρώπη είναι η ελευθερία μας. Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας. Και αυτό που πρέπει να δωρήσουμε στα παιδιά μας είναι ακριβώς αυτό. Ένα μέλλον με ευημερία, με ηρεμία, με ελευθερία.